Mes chers collègues, bonjour. Nous allons... Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Και ε, θα ξεκινήσουμε με το σημείο για την σήμανση και εμπιστοποίηση του ευρωπαϊκού τουρισμού. Ξεκινάμε λοιπόν ε, την απογευματινή συνεδρίαση με την παρουσίαση της μελέτης του Τμήματος Θεματικής Πολιτικής για το θέμα αυτό. Έχουμε την τιμή να έχουμε τους συντάκτες αυτής της έκθεσης μαζί μας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας τους παρουσιάζω πολύ σύντομα. Ο κύριος Richard Βέστον είναι καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο του Κεντρικού Lancashire και ο κύριος Σερμπέρ Αμέν. Είστε πρόεδρος και συνειδητής του ΕΚΟ Trans ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Βιώσιμο Τουρισμό και θα μας παρουσιάσετε αυτή τη μελέτη. Θα είμαι αδιάλακτη ε, επί του χρόνου. Έχετε μόνο 6 λεπτά. Παρακαλώ. Ο κύριος Βέστον έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω τη μελέτη μας. Ο συνάδελφός μου, ο Herbert, θα παρέμβει. Είναι ο αρμόδιος για την βιωσιμότητα, ίσως θέλει να με διορθώσει. Πολύ σύντομη συνόψη λοιπόν. Η μελέτη έγινε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σήματα και πιστοποίησεις και δημιουργούνται με διάφορους τρόπους και οι περισσότεροι πολίτες ε, τους αγνοούν. Είναι πάρα πολλά. Αυτά τα σήματα δεν καταλαβαίνουν σε τι διαφέρουν μεταξύ τους και οδηγεί, οδηγεί και σε σύγχυση τις επιχειρήσεις. Δεν ε, είναι απρόθυμες να επιδιώξουν να λάβουν αυτά τα σήματα. Υπάρχουν περίπου 250 σήματα στην Ευρώπη. 160 από αυτά είναι βιωσιμότητας, 100 περίπου ποιότητας και αυτά είναι σε διεθνέ και εθνικό επίπεδο. Και αν περάσετε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, υπάρχουν ακόμη πολύ περισσότερα. Αυτό δημιουργεί ε, σύγχυση όχι μόνο στου ε, τοπικού τουρίστε, από την ίδια περιοχή δηλαδή, αλλά πολύ περισσότερο από άλλε περιοχέ τη χώρα ή από άλλε χώρε. Ακόμη και ένα από τα σήματα που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, το Q στην ε, Ισπανία για παράδειγμα, μόνο μισό της εκατό των σχετικών επιχειρήσεων το έχουν. Παρά το ότι είναι καθιερωμένο, δεν υπάρχει πολλοί κόσμο να ενδιαφέρεται. Υπάρχει πραγματικά θέμα. Πρέπει να το δούμε. Αυτό εξετάσαμε. Έγιναν ε, κάποιες προσπάθειες να γίνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ήδη δύο μελέτες και προσπάθησαν να εισαγάγουν μερικές αρχές για τον ευρωπαϊκό τουρισμό ποιότητα, αλλά ούτε ένα χρόνο δεν κράτησαν. Υπήρχε μεγάλη αντίσταση από κάποια κράτη-μέλη. Οπότε υπάρχει κάποια ανησυχία για το θέμα της επικουρικότητας. Πρέπει να τα λάβετε υπόψη αυτά τα θέματα, τις απόψεις των ε, ε, ανθρώπων που αμφιβάλλουν. Αλλά σε κάποια κράτη υπήρξε πολύ θετική αντίδραση. Η βιωσιμότητα τα έχει πάει κάπως καλύτερα. Υπάρχει η ενωσιακή, το ενωσιακό σήμα οικολογίας, ε, το οποίο είναι αρκετά αποδεκτό στις χώρες όπου έχει γίνει πολύ παρουσίασή του, πολύ στήριξή του. 5-6 χώρες ε, όπου έχει παρουσιαστεί πολύ και σε αυτές έχει αρκετά μεγάλη διάδοση. Χρειάζεται στήριξη σε εθνικό επίπεδο και παρουσίαση. Πρέπει το κράτος μέλος να σε στηρίζει. Τα άλλα δύο σήματα είναι κυρίως ε, μέσα για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα είναι πιο διαχειριστικά εργαλεία. Ένα από τα κυριότερα μελήματά μας είναι να συζητήσουμε με τους εμπλεκούμενους φορείς, για παράδειγμα με επιμελητήρια, ξενοδοχειακούς ομίλους, άλλες τέτοιες οργανώσεις και τις οργανώσεις που παρέχουν την πιστοποίηση. Όλοι συμφωνούν ότι είναι σημαντικά αυτά τα σήματα για να βελτιωθεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα και βεβαίως για να ενημερώνουν τους καταναλωτές. Έχει λοιπόν διάφορες διαστάσεις. Τα δύο τρίτα των ε, εμπλεκομένων φορέων θεωρούν ότι η ψηλότερου επίπεδου επισημάνσεις ε, λειτουργούν καλύτερα, δηλαδή εθνικού και διεθνού, διεθνούς επίπεδου. Οι οργανισμοί επιστοποίηση είναι κάπως λιγότερο παρεμβατικοί, αυτό δεν θα πρέπει να μα εκπλήσει. Θα ήθελαν περισσότερη στήριξη από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή τα, τα σήματά τους γιατί οτιδήποτε άλλο θεωρούν ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό. Στην ε, μελέτη μας μία σημαντική ψηφία, ένα τέταρτο και πάνω, ήταν κατά της εισαγωγής ε, τέτοιων προδιαγραφών ή σημάτων. Πρέπει να τους πείσουμε και αυτούς, να κατανοήσουν ε, ποια θα είναι τα ωφέλη. Δεν θα είναι απλώς ε, περισσότερη γραφειοκρατία. Εξετάσαμε μια σειρά από περιπτώσεις για να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά σήματα. Αναφέρουμε ορισμένα τα αστέρια για τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα. Αυτό επιβιώνει. Αν και η προσωπική μου γνώμη είναι, είναι ότι είναι πολύ στενό. Κοιτάει μόνο τα δωμάτια και πόσα ξενοδοχεία συμμετέχουν. Δηλαδή δεν επεκτείνεται η χρήση του, απλώς τα αρχικά μέλη και κάποιοι που έχουν προσθεθεί από τη Δανία. Για την, το οικολογικό σήμα το ανέφερα. Τα κριτήρια για τον παγκόσμιο βιώσιμο τουρισμό, GSTC, είναι κάτι που έχει δημιουργήσει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι καλύτερα να απευθυνθείτε σε αυτούς γι' αυτό για να ενημερωθείτε για τα διδάγματα που έχουν αυτοί εξάγει. Το, το σήμα Q επίσης, quality δηλαδή, μοιάζει να ε, ασχολείται με διάφορους τομείς, συγκεκριμένα 23 διαφορετικούς τομείς του τουρισμού και μετά έχουμε τις ε, πλατφόρμες στο ίντερνετ Εδώ προσπαθούν να συνδυάσουν αντικειμενικά κριτήρια με τα υποκειμενικά κριτήρια των ε, απόψεων που εκφράζουν όσοι γράφουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Παρά το ότι μία πρόσφατη μελέτη λέει ότι θα, έπρεπε να είναι δυνατόν να συνδυαστούν αυτά. Αλλά πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Οπότε, συμπεράσματα. Ε, αρκετά προφανή. Αν θέλετε να λειτουργήσει, θα πρέπει να συνδυάζεται με τις άλλες ενωσιακές πολιτικές, να αλληλοϊποστηρίζονται. Να έχετε υπόψη, αν δημιουργήσετε κάτι τέτοιο, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του τουρισμού είναι μικρομεσαίες. Άρα θα είναι πολύ περισσότερη γραφειοκρατία, άρα δεν θα ενταχθούν πολύ εκτός αν τις στηρίξετε πραγματικά, αν είναι επιπλέον αρκετά απλό να εφαρμόσει και να συμμετάσχει κανείς σε ένα τέτοιο σύστημα. Ορισμένες είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δύο-τρεις εργαζόμενοι, δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν ε, το αναγκαίο διοικητικό δυναμικό. Και να δούμε πώς θα μπορέσουν και οι απόψεις που εκφράζουν, οι κριτικές που εκφράζουν στο διαδίκτυο οι πελάτες να ενταχθούν και αυτές σε αυτά τα σήματα. Γιατί υπάρχουν και έχουν σημειώσει αρκετή επιτυχία και έχουν απήχηση στο κοινό με τρόπο που οι παραδοσιακές ε, επισημάνσεις και πιστοποίησεις δεν έχουν. Λοιπόν, γενικά θεωρείται θετική η παρέμβαση της Ένωσης, δεν δημιουργεί επικάλυψη, δεν θα έπρεπε να δημιουργείται επικάλυψη, να μην είναι άλλη μία επισήμανση, δεν θέλουν άλλο ένα σήμα, άλλη μία επιστοποίηση. Πρέπει να είναι κάτι που να βασίζεται σε αυτό που υπάρχει και να το προωθεί, να το ενοποιεί. Ορισμένοι δεν είναι ιδιαίτερα θετικοί. Και αυτό να το λάβετε υπόψη. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση για να ε, ενταχθεί και η ποιότητα και η βιωσιμότητα. Δηλαδή ήδη και κάποια σήματα βιωσιμότητας λαμβάνουν υπόψη κάποια κριτήρια ποιότητας. Κάποια βέβαια ε, όχι. Είναι δύσκολο για πεντάστρα ξενοδοχεία να επιτύχουν και τα κριτήρια βιωσιμότητας γιατί έχουν διαφορετικά κριτήρια. Αλλά εάν ε, θέσετε κάποιους στόχους ε, δεν θα καταλήξετε πουθενά. Συστάσεις. Οι δύο πρώτες είναι πραγματικά να μπορέσουν οι φορείς του τομέα να κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, ακόμη και αυτοί που είναι διστακτικοί, αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν, δεν ενδιαφέρονται, ε, είναι καχύποπτοι όλοι αυτοί από την αρχή να κατανοήσουμε τις ανησυχίες τους, να επιχειρήσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Μόνο έτσι θα πιστούν να συμμετάσχουν σε όλη την πορεία. Όπως είπα, είναι ουσιώδης η μειοψηφία, όπως και για τις προσπάθειες που έκανε προηγουμένως η Κομισιόν. Να μιλήσετε με και το GSTC, που σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και καιρό προσπαθεί να το προωθήσει, να διδαχθούμε από αυτούς, να δούμε αν μπορείτε να συνδυάσετε τις προσπάθειές σας και να είναι απλώς μια ευρωπαϊκή εκδοχή του GSTC. Έχουν ε, εξαγάγει κάποια διδάγματα, έχουν κάνει προσαρμογές. Να μην ε, επανεπινοήσετε τον τροχό. Μιλήστε μαζί τους για να μάθετε από τα διδάγματά του, Να, να ενθαρρύνετε τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού να ε, αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα σήματα για να αυξηθεί η ποιότητα. Υπάρχει μια σκοτσέζικη επισήμανση όπου έκαναν διάφορες προσπάθειες στα ξενοδοχεία, ε, επισκέψεις επιθεωρητών, αλλά οι επιθεωρητές μετά δεν επέκριναν τα ε, ξενοδοχεία, απλώς τους είπαν, κοιτάξτε αυτές είναι οι συστάσεις μας για να βελτιώσετε. Δεν τους είπαν θα σας κόψουμε αστέρια. Τους είπαν θα σας βοηθήσουμε να αυξήσετε την ποιότητα των υπηρεσιών σας. Αυτό ήταν ένα καλό παράδειγμα. Δηλαδή να πείσετε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν με θετική αντιμετώπιση, επικοδομητική. Έχει καλύτερη απήχηση και τοπικέ πρωτοβουλίε βεβαίω. Και το τελευταίο, να το στηρίξετε εσείς οι ίδιοι. Να έχετε πολιτικές που θα λένε εμείς θα χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που να είναι ακριβώς πιστοποιημένες. Έτσι βοηθάτε αυτές τις επιχειρήσεις. Μπορούν να δουν αξία μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμά σας. Έτσι θα σας ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Θα δώσω το λόγο στον συναδελφό σας, τον κύριο Αμέλα. Έχετε 6 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω εκπλαγεί. Δεν ήξερα ότι θα έχω κι εγώ 6 λεπτά, όπως και εσείς. Ωραία. Δεν ήρθα απλά έτσι για να είμαι εδώ. Υπάρχουν 250 σήματα στην Ευρώπη, ορισμένα από αυτά λειτουργούν πάνω από 30 χρόνια και άλλα δημιουργήθηκαν φέτος. Όλα αυτά τα σήματα υποστηρίζονται από πολύ διαφορετικούς ενδιαφερομένους. από κάποιους φορείς, άλλα από τον τομέα της φιλοξενίας, άλλοι από ΜΚΟ, από εθνικές κυβερνήσεις που έχουν υποστηρίξει τη δημιουργία την ανάπτυξη ε, προγραμμάτων πιστοποίηση που τώρα χρειάζεται να ε, επιβιώσουν. Τι σημαίνει αυτό, να επιβιώσουν, να, επιβιώσουν, να έχουν να έχουν αρκετά ξενοδοχεία οι επιχειρήσεις που ετούνται τέτοια πιστοποίηση ως ε, απόδειξη ποιότητας πιστοποίησης πέραν της νομοθεσίας. Αυτό επιζητάει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα με αυτόν τον τρόπο, έστω και ω τάση. Συγκρίνω τη σήματα μαζί με την ομάδα μου εδώ και πάνω από 30 χρόνια και παρατηρώ τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου. κοιτώντα ε, τον διεθνή ανταγωνισμό στον τουριστικό κλάδο, αντιλαμβάνομαι ότι η επισήμανση, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, ε, διαρκώς αυξάνεται ε, και ειδικότερα τα εθνικά γραφεία τουρισμού, από τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού. Στην Γερμανία, ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού πέρυσι ξεκίνησε μια νέα αναγνωρισμένη πρωτοβουλία που ονομάζεται ε, βιώσιμη εμπειρία στη Γερμανία, η γερμανική βιώσιμη εμπειρία, η εμπειρία βιωσιμότητας. Μας ε, ζήτησαν ε, τα στοιχεία και εμείς ε, έχουμε πάει σε πράσινα πιστοποιημένες επιχειρήσεις και προωθούμε παγκοσμίω το, το marketing τους και που αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τους 32 οργανισμούς που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο βλέπουν τα 600 αυτά ξενοδοχεία τα οποία προωθούνται και έχουν, ανήκουν στην κατηγορία της βέσμης ανάπτυξης στη Γερμανία. Βλέπουν και άλλες ε, πρωτοβουλίες. Όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα. Αλλά δεν είναι παρά ένα μόνο παράδειγμα, ένα μόνο πρώτο βήμα. Διότι υπάρχουν και πολλές άλλες επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ε, διάφοροι οργανισμοί δραστηριοτήτων, ε, ταξιδιωτικά πακέτα, ακόμη και προορισμοί που λαμβάνουν πιστοποίηση. Το θέμα είναι τι ε, τους δίνει κάποια ιδιαιτερότητα, για, ποια, που είναι η δύναμή τους, ε, γιατί χαρακτηρίζονται ως κάτι ιδιαίτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, τι χαρακτηριστικά έχουν ποιοτικά βιωσιμότητας ως προορισμοί, τουριστικές υπηρεσίες σε σύγκριση με άλλα αντίστοιχα μέρη υπηρεσίες σε ολοκληρώ τον κόσμο. Και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, αν δείτε τα ελάχιστα περιβαλλοντικά πρότυπα το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα μαζί με το σύστημα διαχείρισης ΣΕΜΑΣ. Ε, τα πρότυπα αυτά είναι παγκοσμίω αναγνωρισμένα και πολύ ψηλά. Ε, δεν έχουν επιτευχθεί σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτή λοιπόν θα μπορούσε να είναι υπερβολητική συνιστόσα για μια σύσταση βιώσιμου τουρισμού ή για μια, ε, ένα σχετικό πρότυπο ε, ένα προσανατολισμό που απορρέει από τα γενικότερα ε, κριτήρια βιωσιμότητα, τα οποία είναι γενικότερα, όπω εφαρμόζονται ειδικότερα στην Ευρώπη και που χρησιμοποιούνται ω σύσταση, ω μηχανισμό επιλογή ε, για όλα εκείνα τα σήματα που δείχνουν ότι στην Ευρώπη είμαστε δυνατοί. Και αυτό βοηθά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορία, τους προορισμούς ε, που λένε ότι από τα 150 περιβαλλοντικά ε, πρότυπα και πρότυπα βιωσιμότητας αυτά τα 20-30 είναι πολύ ε, ισχυρά διότι πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσει σε θέματα περιβαλλοντικά, σε θέματα βιωσιμότητας περιλαμβανομένης της κοινωνική, των κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων είναι κάποια κριτήρια ποιοτικά Κάτι που βοηθά ιδιαίτερα ε, την κατάσταση και ε, που θα χρησιμεύσει σε κάποιες πρόσφατες και σε κάποιες νέες πρωτοβουλίε, τις οποίε δεν συμπεριλάβουμε γιατί ξεκίνησαν μόλις φέτος. Για παράδειγμα, στη Γερμανία υπάρχουν 10.000 ε, ταξιδιωτικά πρακτορία, ω γραφεία φυσικά και οι υπηρεσίε online. Πολλούν κατά κύριο λόγο ταξιδιωτικά πακέτα τουριστικών ε, οργανισμών, τουριστικών φορέων. Το ίδιο βλέπετε και σε άλλες χώρες. Τα ε, συστήματα πληροφοριών αυτών των ταξιδιωτικών γραφείων που ε, όταν κάθεται εκεί ο υπάλληλο μπροστά σε έναν υπολογιστή, συμπεριλαμβάνουν και ένα πράσινο φιλαράκι, το οποίο βασίζεται σε κάποιες βασικές απαιτήσεις. Το ξενοδοχείο, για παράδειγμα, που έχω στο πακέτο μου πρέπει να είναι επιστοποιημένο ε, GSTC, ε, για παράδειγμα, να είναι αναγνωρισμένο από το GSTC το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο στην Ευρώπη. Μετά υπάρχει το Travelport Austria, ένας μεγάλος ανταγωνιστής του συστήματος Bistro, που σχετίστηκε με το, συνδέεται με τον Galileo κτλ. Αυτοί λένε ότι δεν, είναι, δεν υπάρχει μόνο αναγνώριση GSTC αλλά και EU ECO και άλλα συστήματα πιστοποίησης έχουν πολύ ψηλή ποιότητα ειδικότερα σε περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία ε, είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη. Θέλουμε να προωθήσουμε και αυτά. Και τα δύο και πολλά άλλα συστήματα όπως και υπηρεσίες κρατήσεων όπως ε, ε, η ECO BNB για παράδειγμα, όχι Airbnb χρειάζονται κάποιο είδου ευρωπαϊκή καθοδήγηση. Ε, από όσο καταλαβαίνουμε εμεί από τα σχόλια που έχουμε λάβει ε, για τις διάφορε μελέτε. Το τελευταίο που ήθελα, ήθελα να αναφέρω είναι ότι όλα αυτά είναι εφικτά, αλλά χωρίς να ξεχνάμε τα υπάρχοντα σήματα, τα οποία λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό, ε, εθνικό και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εμπειρία από αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των προτύπων στην Ευρώπη συνολικά, ώστε να καταλήξουμε σε μια ε, πολύ καλή ποικιλία ε, και πολυμορφία σημάτων για την, βιωσιμότητα, για την ποιότητα όπως καθορίζεται από τους ε, πελάτες. Και είμαι σίγουρος ότι θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αμέλ. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Βαντεκάμ. Επιτρέψτε μου απλώς να πω ότι... Συγγνώμη, Κλάδιο Μοντέρο και Λουίντε Μπόρντες. Από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ως τουριστικοί οι δήμονες. Απολογούμε λοιπόν για την απουσία τους. Επιτρέψτε μου απλώς να ευχαριστήσω τον κύριο Χάμελα και τον κύριο Βέστερν για την έκθεσή τους που μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για όλα όσα συμβαίνουν στον τομέα αυτό. Και είναι αρκετά παρατηρητική. Στις διακοπές μου μου έκαναν πολλές ερωτήσεις. Γιατί, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ένα σύστημα επισήμανσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον τουρισμό. Και είναι μια ολόκληρη συζήτηση σχετικά με το ποια, ποιοι είναι η βασική στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό... Και αυτή είναι η ερώτησή μου για τον κύριο Βέστεν. Είναι λογικό για την Επιτροπή να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τις τουριστικές επισημάνσεις μήπως θα ασχολείται με λεπτομερή πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο ΕΠΠ σε ό,τι αφορά τα σήματα, τα ταξιδιωτικά σήματα. Σε ό,τι αφορά τα σήματα στους, στους δρόμους. Αν έχουμε την επιλογή θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα μεγάλα ζητήματα. Εγώ προσωπικά μου αρέσει πολύ το TripAdvisor σαν μηχανή αναζήτησης, αλλά δεν πηγαίνω ποτέ εκεί για να βρω ξενοδοχείο, για παράδειγμα. Πολύ συχνά εκεί πηγαίνουν γκρουπ Κινέζων. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους ε, Κινέζους τουρίστες, αλλά είναι μεγάλα νούμερα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον οδηγό Michelin, οποιοδήποτε ψάχνει για καλό φαγητό μπορεί να ακολουθήσει τον οδηγό Michelin. Γιατί δεν υπάρχει κάτι ανάλογο και στον τομέα του τουρισμού. Με άλλα λόγια, μου αρέσει η έκθεση αυτή γιατί μας δίνει μια γενική εικόνα της κατάστασης δεν θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις νεόφυτες επιχειρήσεις, δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις για αυτές τις νέες επιχειρήσεις, αυτού του τύπου οι λίστες. Και πώς κανείς μπορεί να μπει σε αυτές τις λίστες. Αυτά είναι δύο μικρά ζητηματάκια Και πάλι, όπως είπα, δεν θεωρώ ότι αφορούν την Ευρώπη εν γέννη. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ντεμόντε και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολλές φορές ε, θεωρούμε ότι δεν δίνεται επαρκής προσοχή στον τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευπρόσδεκτες λοιπόν όλες οι πρωτοβουλίες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και να αποτελέσουν κίνητρα ε, για την αύξηση περισσότερων τουριστών και για τη βελτίωση της ποιότητας. Όσον αφορά την επισήμανση, είναι πολλές, ε, ε, πολλά τα σήματα, ίσως υπερβολικά πολλά. Καλό θα ήταν να υπάρξει κάποια ρύθμιση, κάποια εναρμόνιση. Αυτό θα βοηθήσει να είμαστε και πιο σαφείς προς τους τουριστές που έρχονται ε, από χώρες εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί σε διεθνές επίπεδο πιστεύω είναι ακόμα πιο ασαφής αυτή η σήμανση. Δύο θέματα ήθελα να αναφέρω, ε, δύο ερωτήσεις. Ε, η πρώτη αφορά την ταυτοποίηση. Καθώς εσείς μιλούσατε, εγώ προσπάθησα να κάνω μια έρευνα μέσω μιας γνωστής πλατφόρμας για να δω κατά πόσο αναφέρεται πιθανά αυτού του είδους η σήμανση. Δεν αναφέρεται. Ακόμη και αν αναζητήσει κανείς τα κριτήρια, τα διάφορα κριτήρια προσφοράς ε, υπηρεσιών δεν υπάρχουν πουθενά τέτοια σήματα. Εσείς προηγουμένως αναφερθήκατε σε τουροπερέτες, σε διαργωνωτές ταξιδιών και σε πρακτόρια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, το 95% των τουριστών ε, κάνουν αναζήτηση μέσω πλατφορμών. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ψηφιακά συστήματα. Η επιλογή δηλαδή θα πρέπει να γίνεται ε, στην αρχή της έρευνας, όχι αφού φτάσει ο τουρίστας στον προορισμό του. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξή. Πώ θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τη συμμετοχή αυτών των ψηφιακών φορέων ώστε ε, να προωθηθεί μέσω τη ψηφιακή τεχνολογία η σήμανση αυτή και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η δεύτερη μου ερώτηση. η ανακοίνωση για περιβαλλοντικά θέματα σε διάφορα ξενοδοχεία γίνεται περισσότερο ε, για, με σκοπό τιμή των ε, δαπανών τους. Ουδέποτε έχω δει να γίνεται διαλογή απορριμμάτων σε ε, ξενοδοχεία. Ο κάθε τουρίστας παίρνει μαζί του τις διάφορες συνήθειες που έχει στο σπίτι του. Ε, και στις διακοπέ του όσον αφορά τη διαλογή των απορριμμάτων. Ε, τι διαδικασίες λοιπόν θα μπορούσαν να ακολουθηθούν για να έχουμε μείωση των απορριμμάτων, για τη διαλογή των απορριμμάτων. Ε, χαίρομαι λοιπόν για τον αριθμό των σημαντών που έχετε συμπεριλάβει και τον αριθμό των ενδιαφερομένων και εγώ βλέπω πολλούς ενδιαφερομένους από την Ιταλία από τη χώρα μου, αλλά γιατί να μην έχουμε και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που είναι ειδικευμένε στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση, στη διάδοση των γνώσεων για θέματα ε, που αφορούν ακριβώς αυτές τις ε, τουριστικές υπηρεσίες με σεβασμό προς το περιβάλλον. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε, κυρία Φώστερ, έχετε λόγο. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που έχασα τα αναρτήρια σχόλια, αλλά σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπεριστατωμένη έκθεση που μας παρουσιάσετε. Εγώ εργαζόμουν στην τουριστική βιομηχανία, στην βιομηχανία αερομεταφορών και γνωρίζω τα ζητήματα που αφορούν στη συμμόρφωση των ξενοδοχείων και πιστεύω ότι κανένας μας βασικά δεν είναι ενάντια στην επισήμανση, στα σήματα που χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο, με τους σωστούς δείκτες δηλαδή δεν έχει να κάνει με το πόσες ετικέτες έχουμε, έχει να κάνει με το πώς συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις με τις ετικέτες αυτές. Δηλαδή μπορεί να αποκτήσουν την ετικέτα, την επισήμανση, τη διαπίστευση και μετά να μην συμμορφωθούν ένα-δύο χρόνια, μετά να μην συμμορφώνονται. Θεωρώ ότι εκεί έγκυται το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της βιωσιμότητας, τα σήματα βιωσιμότητας, το υποστηρίζω 100% και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο οι τουριστικοί πράκτορες αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες είναι κάτι το οποίο λαμβάνουν υπόψη τους αλλά και οι καταναλωτές ε, τι περιμένουν να δουν δηλαδή με άλλα λόγια όταν πηγαίνουν σε ένα μέρος ή όχι. Για μένα κάποια από τα βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές είναι ότι δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει να σταματάμε καταρχήν στα σύνορα των κρατών μελών αλλά κοιτάζουμε την Ευρώπη στο σύνολό τη. Αυτό που θα πρέπει να εξετάζουμε είναι κατά πόσο ένα τετράστορο ξενοδοχείο είναι ένα πραγματικά ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Δηλαδή σε μια χώρα ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων είναι το αντίστοιχο ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων σε κάποια άλλη χώρα. Είναι κάπως σχετικό το να, να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα, τα αστέρια σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία. Τι ακριβώς μας δίνει να καταλάβουμε το κάθε σήμα. Κάποια άλλα βασικά ζητήματα για το κοινό οποιοδήποτε ξενοδοχείο πηγαίνουν ή οποιοδήποτε bed and breakfast θα πρέπει να προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι πρόκειται για ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν ζητήματα, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το φαγητό που προσφέρεται. Είναι ένα αβαντάζ για τον καταναλωτή να ψάχνει, να γνωρίζει πού πηγαίνει. Είναι οι ίδιοι βέβαια υπεύθυνοι για τις επιλογές όταν πηγαίνουν σε διαφορετικά κλίματα, για παράδειγμα. Το τελικό ζήτημα που θέλω να θέσω είναι ότι όταν εξετάζουμε τα σήματα σε ό,τι αφορά ε, One of the biggest Ένα από τα βασικά ζητήματα έχει να κάνει με, την, ε, με τα άγρια για παράδειγμα. Όλα και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται να πάνε σε σε μέρη που αντιμετωπίζουν τη, τα άγρια ζώα με, έναν, με σεβασμό. Δεν ε, πηγαίνουν σε χώρες που δεν σέβονται κάποιους γενικούς κανόνες, για παράδειγμα τα, για τα δέσποτα ζώα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, γιατί αν κοιτάξουμε την ατζέντα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζώων, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται παντού. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα για την εταιρεία Emirates, για παράδειγμα, την αεροπορική εταιρεία. Σε ό,τι αφορά τον Αφρικανικό ελέφαντα, η ίδια η βιομηχανία προσπαθεί να προωθήσει αυτή την ιδέα της βιωσιμότητας σε κάποιες περιοχές, να προωθήσει περιοχές όπου οι ίδιες οι χώρες αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί για τον ε, πληθυσμό των ζώων που βρίσκονται εκεί. Είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές που έχουμε θέσει σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ζώων για τα οποία μαχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απλά ένα ζήτημα που ήθελα εγώ να θέσω, γιατί θα ήθελα να δω να γίνεται αναφορά σε αυτό το ζήτημα γιατί πιστεύω ότι γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Έχουμε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη βιομηχανία εδώ στην Ευρώπη. Πιστεύω, θεωρώ ότι έχουμε να προσφέρουμε πολλά στου ανθρώπου που έρχονται από όλο τον κόσμο, αλλά βεβαίω μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Σα ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε κύριε Φώστερ. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για τη μελέτη. Σημαντικά πράγματα μας είπατε Έχουμε πάνω από 250 σήματα, οπότε τίθεται το ερώτημα. Τι κάνουν ε, οι διάφοροι μπλεκόμενοι του κλάδου. Ε, τι κάνουν οι καταναλωτές. Εγώ δεν ε, πρόκειται να κοιτάξω 250 σήματα για να διαπιστώσω ποιο έχει έννοια και ποιο δεν έχει. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Πώς τα αντιμετωπίζουν ο κλάδο επιχειρεί, δηλαδή να υπάρξει κάποια απλούστευση, κάποια ενοποίηση. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχο μα. Πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιε δικέ μα προδιαγραφέ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση. Αν δεν υπάρχει, δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο, ούτω ώστε να ικανοποιηθούν και οι επιχειρήσει και οι πελάτε. Πώς μπορεί δηλαδή η Ένωση να συνεργαστεί επιτυχώς προς αυτή την κατεύθυνση και με τις εθνικές αρχές. Να σας ε, δώσω ένα παράδειγμα από εντελώς άλλο τομέα. Όπως ξέρετε, ε, έκανα αποδηλασία σε μια ε, συγκεκριμένη διαδρομή που λέγεται Ευρωπαϊκό Κύμα. Είχα πάει, στην, για παράδειγμα, συγκεκριμένα στο Κόλοπτσεκ, στην ακτή της Πολωνίας υπήρχε εκεί ένας θαυμάσιος ποδηλατόδρομος και ένα τεράστιο σήμα που έλεγε συγχρηματοδοτήθηκε ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε ορισμένα άλλα σημεία αυτής της ε, διαδρομής δεν υπήρχαν σήματα. Αναφερόταν απλώς ένα σήμα R1, το οποίο πρέπει να ρωτήσεις, όπως ρώτησα και εγώ. Ενώ χρηματοδοτούμε δεν υπάρχουν σήματα, δεν υπάρχουν πινακίδες που να τα λένε. Πήγα στη Ρουμανία, κατά μήκο του Δούναβη θαυμάσιες πινακίδες και για τα ε, για παράδειγμα τους αρχαιολογικούς χώρους αλλά μόνο στα ρουμάνικα έλεγε βεβαίως συγχρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εγώ δεν ξέρω ρουμάνικα και πολλοί άλλοι δεν ξέρουν ρουμάνικα αλλά θα ήθελα να έχω λάβει αυτή την πληροφόρηση πως είναι δυνατόν να αποδέχεται η Κομισιόν ότι χρηματοδοτεί τόσα πράγματα χωρίς να το μαθαίνει κανείς δεν περίμενα να υπάρχει στα γερμανικά, αλλά τουλάχιστον στα αγγλικά και στην ε, Τσεχία. Ναι, βεβαίως. Έκανα ε, ποδηλασία κατά μήκο του Έλβα. Και πάλι εκεί υπήρχαν πινακίδες, αλλά τίποτα στα ε, αγγλικά. Αλλά στη Σερβία Υπάρχει ε, ο Ευρωπαϊκός Δρόμος 13 ε, που είναι ε, πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα κατά μήκος του Δούναβη. Είναι η λιγόμενη διαδρομή του σιδηρού παραπετάσματος και είναι 720 χιλιόμετρα της Ευρωπαϊκής Οδού 13 όπου αναφέρονται όλα στα αγγλικά και στα αγγλικά η Σερβία που δεν ανήκει είναι αξιοσημείωτο παράδειγμα προς ε, αντιγραφή. Έθεσα λοιπόν μετά από αυτά που είδα στην Πολωνία ένα ερώτημα και τους λέω μα δεν σας πειράζει, δεν σας πειράζει. Το βασικό είναι να τους δώσετε τα λεφτά και τα κράτη και οι οργανισμοί. Δεν θα το σκεφτούν αυτοί, αυτοί έχουν πάρει τα λεφτά. Αν θέλουμε να έχουμε υπόψη τους καταναλωτές και τους ε, διοργανωτές ταξιδίων πρέπει να θέσουν προδιαγραφές. Είμαι πεπισμένος ότι εάν ε, ε, διαπίστωναν όλοι ότι όλα αυτά τα διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα μιμούνταν το παράδειγμά μας και άλλες χώρες. Έτσι θα υιοθετεί το κάτι τέτοιο παγκόσμια. Πιστεύω ότι ορισμένοι λένε ότι είναι κατά. Είναι θέμα ε, εθνικών εγωισμών. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν έχουμε αυτές τις προδιαγραφές θα υποφεληθούμε όλοι οικονομικά θα ήταν ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την κατάσταση, ένας μοχλός. Γι' αυτό σα θέτω σε εσά το ερώτημα πώ μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά και προ την Κομισιόν, γιατί το ανέχετε τόσα χρόνια, ίσω δεκαετίε. Γιατί δεν αναλαμβάνετε κάποια πρωτοβουλία να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να πείτε θα πάρετε μόνο τα λεφτά για τον ποδηλατόδρομο, για τον ευρωπαϊκό δρόμο κτλ. Έχουμε 15 ε, τέτοιου δρόμου, πάνω από 17.000 χιλιόμετρα. Θα τα λάβετε μόνο εάν υπάρχει πινακίδα που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό σήμα. Δεν χρειάζεται να ξαναβρούμε τίποτα καινούριο, να εφαρμόσουμε μόνο αυτά που υπάρχουν. Ευχαριστούμε, πολύ, κύριε Κράμερ. Είχα και δικό δύο ερωτησούλες. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για σήματα και για βιωσιμότητα. Τι σημαίνει βιωσιμότητα? Ποια είναι τα κριτήρια? Κρατάει κανείς κάποιο χάρτη και υπολογίζει ε, κατά τη διαδρομή του πόσα εκπομπέ εκπομπές ας πούμε καυσαερίων ε, εξέπεψε κατά τις διακοπές του. Αυτός είναι ο υπεύθυνο τουρισμός, η ευαισθητοποίηση του καθενός από εμάς. Πώς χαρακτηρίζεται η βιωσιμότητα, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια και σε τι βασίζεται. Λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρο την ε, τουριστική αλυσίδα, η κυρία Ντεμόντε. Μιλήσατε για τα ξενοδοχεία και τα λοιπά, αλλά οι μεταφορές που πήγαν. Και η τοπική διάσταση βιώσιμος τουρισμός σημαίνει τοπικός τουρισμός που αξιοποιεί την τοπική διάσταση. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να δούμε μαζί ας ε, κάνουμε μια προβολή προς το μέλλον. Βάσει της μελέτης σας, πώς βλέπετε το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού. Κατά την άποψή σας, ως εμπειρογνώμονες, ε, Ποιε θεωρείτε ότι είναι οι πιθανές οδοί για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού. Τι είναι βιώσιμος τουρισμός κατά την άποψή σας. Όλοι λένε θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σήμα. Ναι, πολύ ωραία. Αλλά η σύγκριση με τον οδηγό Μισλά του Βιμ Βαντεκάμπ, ξέρετε εμένα Βιμ Βαντεκάμπ, μα τρελαίνομαι να τρώω, μου αρέσει πάρα πολύ. Το ξέρετε, πώς το ξέρετε. Αλλά όταν πάω και βλέπω τον, τους οδηγούς Μισλά, η, τα κριτήρια είναι κάποια αστεράκια τα οποία τα δίνει ποιο. Ποιο συντάσσει, ποιο ε, ποιος αποφασίζει ποιοι είναι οι εμπειρογνώμονε του οδηγού Μισλά. Γιατί είναι εμπειρογνώμονε, είναι ειδικοί είναι παλιοί σεφ δηλαδή οι οποίοι δίνουν τα αστέρια αυτοί. Όταν έχει κάποιο τρία αστέρια δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πάει να φάει κανεί αυτόν. Ε, αν έχει ένα μόλις ξεκινάει αλλά εκεί είναι το ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα παρέχουν αυτά τα σήματα. Βάσει ποιου εργαλείου, ποιο όργανο θα παρέχει τέτοια σήμα. Αυτό θα ήθελα να γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, έχετε ο καθένας σας 3 λεπτά και 47 για να απαντήσετε. Ακριβώς. 4 λεπτά σας δίνω. άντε 4. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιος ξεκινάει, κύριε Weston. Κύριε Άμελε, ξεκινήστε. To keep a story short. Για να μην μακρηγορώ. Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του να συνδυάζουμε στο έπακρο της προσδοκής ποιότητας και βιωσιμότητας. Την ποιότητα την ορίζουν οι πελάτες. Οι πελάτες είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων σε κάποιον τουριστικό προορισμό που έχουν άλλες απαιτήσει ποιότητας, ε, για παράδειγμα λόγω της ηλικία τους από μια ομάδα πιο μεγάλη ηλικία ανθρώπων που αναζητούν κάποιο πιο ήρεμο μέρος. Αυτή είναι μία μονοπτυχή που μας ε, αποδεικνύει ότι την ποιότητα την καθορίζουν οι πελάτες, ενώ τη βιωσιμότητα δεν την καθορίζουν οι πελάτες. Τη βιωσιμότητα την καθορίζουν τα Ηνωμένα Έθνη με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ειδικότερα όσον αφορά τον τουρισμό. Έχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη στο στόχο 12, την βιώσιμη παραγωγή και εκεί η επισήμανση είναι ένα βασικό εργαλείο για όσους έχουν την αρμοδιότητα για προϊόντα, για τη διανομή τους, για την κατανάλωση. Η κατανάλωση ε, επίσης ε, ενέχει ευθύνη. Ε, εκεί όμως πρέπει ακριβώς να υπάρχουν οι πληροφορίες, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες να λαμβάνονται υπόψη, να μεταφέρονται και να προβάλλονται με τρόπο κατανοητό και ελκυστικό. Και εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει ένα σωρό πράγματα χωρίς όμως να υπάρχει μια ευρωπαϊκή καθοδήγηση. Δεν χρειάζεται να, αντικαταστήσουμε τα σήματά τους. Τα σήματά τους είναι ήδη καθιερωμένα και αναγνωρισμένα. Χρειάζονται όμως μια ευρωπαϊκή καθοδήγηση, έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε τώρα όσον αφορά τι διάφορε ερωτήσει, αλλά θα έλεγα το εξή. Η εξοπιστία των σημάτων. Η κυρία Φώστερα ανέφερε την εξοπιστία των σημάτων, νομίζω. Φυσικά, αν δει τα 150 ε, σήματα για την περιβαλλοντική απόδοση και, την και τη βιωσιμότητα όχι μόνο για, τα, ε, για τις υπηρεσίες φιλοξενίες αλλά και για τα εστιατόρια, για τα αξιοθέατα, για ολόκληρη ουσιαστικά την αλυσίδα ε, υπηρεσιών έχετε σήματα με, βασισμένα σε άριστα πρότυπα αλλά ίσως όχι στα καλύτερα συστήματα επαλήθευσης. Τι σημαίνει αυτό ότι η αξιοπιστία είναι εξίσου σημαντική με την υποσχόμενη ε, βιωσιμότητα. Τι κάναμε λοιπόν πρόσφατα πριν λίγους μήνες, δημοσιεύσαμε με συγχρηματοδότηση μάλιστα του Erasmus Plus, του Knowledge Alliance Program, ε, δημοσιεύσαμε έναν μηχανισμό γρήγορης έβρεσης ε, πιστοποίησης, ώστε εγώ ως ξενοδοχείο, ως υπηρεσία μεταφορών, ως αξιοθέατο να πηγαίνω και να ψάχνω να βλέπω ε, τα συστήματα πιστοποίησης ε, της αναγνώρισης GSTC και να βρίσκω τι υπάρχει και να κάνω ένα κλικ πάνω στο σήμα, να βλέπω ποια είναι η διαφορά και ακόμα καλύτερα ως ε, tour operator να πηγαίνω να κάνω ένα κλικ σε ένα κουμπί ενός χάρτη για να βρω τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις για τους διαχειριστές συγκεκριμένων προορισμών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν ποια ξενοδοχεία, ποιες επιχειρήσεις μας έχουν πιστοποίηση με οποιοδήποτε σήμα. Σήμερα όμως με αυτό το σύστημα μπορούν να πάνε να δουν και να βρουν ότι ένας προορισμός σε σχέση με άλλους προορισμούς είναι λίγο αδύναμος ε, και να δουν πώς κατάφερε ο τάδε προορισμός να έχει 36 ας πούμε επιχειρήσεις στο δρυμό ενώ στον Φραγκενβάλντ έχουμε μόνο 6 για παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αιτίε λοιπόν, οπότε να, οι αιτίες αυτές να αφορούν την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και έτσι να λάβουν κάποια υποστήριξη και να πούν «Α, να, εδώ βλέπω κάτι το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα, ας ε, το υποβάλλω στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Γερμανίας για να το συμπεριλάβει στη γενική του παρουσίαση». Το ίδιο και σε άλλες χώρες Αν δούμε διεθνεί οδού, ε, για παράδειγμα ε, ε, διεθνείς ποδηλατοδρόμους, υπάρχει συγκεκριμένη ποιότητα. Οι, οδές, οι οδοί αυτές μπορούν να αποτελέσουν πρεσβευτή του βιώσιμου περιβαλλοντικού τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά ο τουρισμό δεν σταματάει στα σύνορα, ούτε στα σύνορα των κρατών μελών. Δείτε τη Σερβία. Δείτε λοιπόν όλα τα προγράμματα και τα ε, προγράμματα που λαμβάνουν υποστήριξη με ευρωπαϊκά χρήματα. Ε, εκεί θα βρείτε πολλές καλές πρακτικές που θα έλεγα μπορούν να μας δώσουν πολλές καλές ιδέες και ευκαιρίες για να ε, φέρουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Βουέστα. Να έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εντάχει. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο ερώτημα, κατά πόσο θα πρέπει να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι υπάρχουν ισχυρές απόψεις. Ως επιστήμονας, όταν ξεκίνησα την έρευνα αυτή, προσπάθησα να έχω ένα ουδέτερο, να έχω μια ουδέτερη οπτική γωνία. Να ψάξουμε, να μάθουμε, να βρούμε. Και το ερώτημα είναι απλό το παρόν σύστημα λειτουργεί, το παρόν σύστημα πιστοποίησης. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανώς όχι, είναι, διαφοροποιείται πάρα πολύ. Κάτι το οποίο θίγει την αξιοπιστία του. Κάποια από τα σήματα είναι απλώς αιτήσει που κάποιος πρέπει να συμπληρώσει και παίρνει το σήμα. Επομένως, όχι, το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί. Το δεύτερο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε εμεί να κάνουμε κάτι για να το βελτιώσουμε ή αν θα χειροτερέψουμε τα πράγματα. Και μόνο αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό θα πρέπει να είναι ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα πάντοτε. Κατά πόσο βελτιώνουμε την κατάσταση. Αν θεωρούμε ότι βελτιώνουμε την κατάσταση, τότε καλώ βαίνουμε. Διαφορετικά θα πρέπει απλά να αποδεχτούμε την ήττα μας και να αποσυρθούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσετε. Η γνώμη μου ως οικονομολόγος είναι ότι το υπάρχον σύστημα ε, προκαλεί μεγάλη βεβαιότητα στους καταναλωτές και η αβεβαιότητα στους καταναλωτές και στους ανθρώπους γενικότερα αποτελεί εμπόδιο στο να κάνει κανείς κάτι. Είχαμε μια συζήτηση μόλις πριν έρθουμε. Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς όταν πηγαίνουν για κάπου διακοπέ είναι επειδή δεν καταλαβαίνουν το σύστημα. Θα πρέπει να αγοράσει τα εισιτήρια από πριν, θα πρέπει να πληρώσει μετά, θα πρέπει να έχει μια κάρτα. Δεν ξέρουν πώς ακριβώς λειτουργεί το κάθε σύστημα. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουν όλες αυτές οι διαφορετικές, τα διαφορετικά σήματα είναι κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα στους καταναλωτές και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει, θεωρώ. Μόνο όμως αν πιστεύετε ότι μπορείτε να το καλυτερεύσετε. Και αυτό πιστεύω μας οδηγεί και στα ζητήματα βιωσιμότητας. Είναι τρεις τομείς βιωσιμότητας. Πρώτα απ' όλα το περιβάλλον, η οικονομική βιωσιμότητα και η κοινωνική βιωσιμότητα. Και αν αυτά τα τρία ζητήματα δεν εξισορροπούνται, τότε όλα είναι μάταια. Αν δεν μπορέσουμε να φροντίσουμε το περιβάλλον, δεν έχουμε που να ζήσουμε. Αν δηλαδή επιχειρήσεις τα πάνε καλά, αλλά καταστρέφουν το περιβάλλον, τότε ποιο το νόημα, γιατί να ενθαρρύνουμε τον τουρισμό, όπως συμβαίνει σε κάποια σημεία της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου όταν ο τουρισμός βλάπτει την περιοχή. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να εξισορροπούνται. Αυτή είναι η ουσία της βιωσιμότητας, να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Όλοι πρέπει να δουλέψουμε, όλοι πρέπει να φάμε, πρέπει να υπάρχουν δουλειές, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και για το μέλλον, πρέπει να φροντίσουμε για το περιβάλλον. Πρέπει να στηρίξουμε τις κοινωνικές δομές. Είναι ένα ζήτημα ισορροπίας λοιπόν. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά. Ευχαριστούμε. Κυρία Μέλ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ξέχασα να αναφερθώ σε μια πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή των βιώσιμων στόχων σε 200 περίπου κράτη-μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες του ΩΣΑ, κάτι που αφορά την Ευρώπη και ιδίως την Δυτική Ευρώπη. Τα πορίσματα δείχνουν ότι οι χώρες του ΩΣΑ είτε έχουν αποτύχει, είτε δείχνουν ότι θα αποτύχουν σε ορισμένους στόχους, συγκεκριμένα τους στόχους 20-30, 20 μέχρι 30. Επίσης, ό,τι αφορά το στόχο 12, για τη βιώσιμη κατανάλωση, για την βιοπικιλότητα στην στεριά και στη θάλασσα, αλλά και τον τέταρτο στόχο σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, προσαρμογή και αντιμετώπιση. και οι στόχοι αυτοί αφορούν και αρκετά κριτήρια που μπορείτε να βρείτε σε σήματα σε βιωσιμότητας και σε επιστοποιημένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Είναι μόλις το 1%, θα μπορούσε όμως να φτάσει το 10% ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών. Αν εξετάσουμε όλες αυτές τις εταιρείες που για παράδειγμα δεν ετούνται καν να αποκτήσουν τα σήματα αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο. Αυτός είναι ένας άλλος πολύ ισχυρός λόγος να στηρίξουμε τον τουρισμό ως ε, μοχλό της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε. Αλλά τώρα να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε ε, διάθεση να μας πείτε κάτι. Τρία λεπτά παρακαλώ. Τρία λεπτά. Ο χρόνος έχει ήδη ξεκινήσει να μετράει. Παρακαλώ. Η παρουσίαση της μελέτης κατέδειξε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Κατανοούμε και εμείς την πολυπλοκότητα. Όπως αναφέρθηκε, η Κομισιόν το 2014 υπέβαλε μια πρόταση για μια σειρά εθελοντικών κριτηρίων για ε, τους χώρους ε, διαμονής. Αλλά η πρόταση αυτή δεν προχώρησε για λόγους επικουρικότητας και για λόγους έλλειψης ε, σαφούς προστιθέμενη αξία. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα του τουρισμού για να φτάσουμε σε μια πιστοποίηση ευρωπαϊκού επίπεδου. Πρέπει να δράσει κανεί πολύ προσεκτικά και πολύ εμπεριστατωμένα. Διότι οι τουριστικές υπηρεσίες ε, είναι πολύ διαφορετικέ. Και χρειαστήκαμε πολύ χρόνο για να ζητήσουμε τι σημαίνει διαμονή και ξενοδοχεία Αναφέρθηκαν και τα εστιατόρια φυσικά. Και υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο τουρισμός. Είναι δύσκολο λοιπόν να τις ε, καθορίσουμε. Και πρέπει παρόλα αυτά να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Υπάρχουν μια σειρά από ε, προσπάθειες πιστοποίησης. Η Κομισιόν το παρακολουθεί από πλευράς ε, βιωσιμότητας του τουρισμού, ενθαρρύνει τον κλάδο να εφαρμόσει μέτρα αυτορύθμισης. Ξέρουμε ότι τα ξενοδοχεία και τους χώρους διαμονής ε, γενικά λειτουργεί αρκετά καλά. Ή να συμμετάσχουν σε τέτοια σήματα εθνικά ή περιφερειακά που ήδη λειτουργούν. Λάβαμε τη μελέτη, θα μελετήσουμε τις συστάσεις, θα δούμε τι είναι εφικτό στα πλαίσια των περιορισμένων αρμοδιοτήτων μας για τουριστική πολιτική, αλλά αφορούν και τον ίδιο τον κλάδο, τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και τον, ε, τις εθνικές ε, αρχές τα θέματα αυτά. Να απαντήσω στον κύριο Κράμερ. Αναφερθήκατε στα, ε, στους ποδηλατοδρόμους Eurovelo που ε, διαχειριζόμεθα στην Ευρώπη. Όλα όσα χρηματοδοτούμε πρέπει να ε, αφορούν, πρέπει να συμμορφούνται με τις προδιαγραφές ε, του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα εξετάσω λοιπόν τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες συμβάσεις για να δω τι προέβλεπαν για τη σήμανση και θα σας ε, στείλω απαντήσεις. Θίξατε λοιπόν ένα θέμα για το κατά πόσο θα πρέπει ε, τα σήματα αυτά να λαμβάνουν υπόψη το ότι υπάρχουν και ξένοι τουρίστες που κάνουν ποδήλατο σε αυτούς τους διαδρόμους και θα επανέλθω λοιπόν αφού το εξετάσω. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Κυρία Θαλασσοπούλου. Ε, μακροσκελές το επίθετό σας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, ευχαριστώ κύριε Βέστον και κύριε Αμέλ για την παρουσίαση της εκθεσής σας και πάντα θα είστε καλοδεχούμενοι στην Επιτροπή μας. Θα τα πούμε λοιπόν και θα ε, επιδιώξουμε να παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό για να υπάρξει μια εναρμόνιση ούτως ώστε να μην είναι φραγμός αλλά αντίθετα να είναι μια ευχάριστη δυνατότητα για τους ε, πελάτες, για τους ταξιδιώτες να μπορέσουν να διαλέξουν καλύτερα να τους χειροκροτήσουμε. Και συνεχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι τις εργασίες μας. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που αφορά το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη για την έρευνα και την καινοτομία. Θα συζητήσουμε τις δύο γνωμοδοτήσεις. Τη μία αφορά την πρόταση κανονισμού για την λειτουργία του προγράμματος Ορίζον Ευρώπη και το άλλο αφορά την απόφαση των ειδικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα για τις μεταφορές. Και να δώσω απευθεία το λόγο στην κυρία Βίρκουνεν για να μας παρουσιάσει τα σχέδια γνωμοδότηση που θα αποστείλουμε στην Επιτροπή Ήτρε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Horizon Ευρώπη είναι ένα πακέτο, αλλά έχει δύο τμήματα. Είναι ο κανονισμός και υπάρχει και μία απόφαση. Αλλά είναι ένα ενίο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό, Horizon Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον μας. Το, πρόγραμμα, το πρόβλημα που υπάρχει τώρα με το Horizon 2020 είναι ότι ήταν τόσο επιτυχημένο, τόσο δημοφιλές, που μόνο 12% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έλαβαν χρηματοδότηση. Άρα έχουμε μεγάλο θέμα, γιατί υπευλήθησαν ε, πολλές ε, προτάσεις ε, υψηλής ποιότητας και πολλές από αυτές δεν στηρίχθηκαν. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο επιμένει ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού κατά την επόμενη περίοδο και με αυτό συμφωνεί και η Κομισιόν. Και για τη δική μας Επιτροπή είναι σημαντικό να στηρίξουμε αυτή τη γραμμή. Την άνοιξη το Κοινοβούλιο πρότεινε μια αύξηση κατά 50% του προπολογισμού του προγράμματος αυτού όταν ψηφίσαμε στην Ολομέλεια. Η Επιτροπή προτείνει αύξηση αλλά όχι τόσο σημαντική. Γι' αυτό προτείνω στη γνωμοδότησή μας να τονίσουμε ότι θέλουμε 50% αύξηση. Αυτή ήταν η άποψη του Κοινοβουλίου, όπως ενεκρίθη από την Ολομέλεια την Άνοιξη. Δηλαδή άνω των 131 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινέ τιμέ. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα από τα κύρια μηνύματα που πρέπει να αποστείλει η Επιτροπή μα, γιατί ξέρουμε ότι είναι ζωτική σημασία για το μέλλον μα. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Συνολικά νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι αρκετά ισορροπημένη και σκόπιμη. Η Κομισιόν λέει ότι το νέο πρόγραμμα θα είναι εξέλιξη, όχι επανάσταση προτείνει μερικά νέα στοιχεία, να έχουμε μια πιο στόχο προσιλωμένη προσέγγιση και νέους προσανατολισμούς για τον προπολογισμό για την ε, άμυνα. Καλύπτει το πρόγραμμα πολλούς σημαντικούς τομείς των μεταφορών, ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση, ασφάλεια και φυσικά κατάργηση των εκπομπών ε, οξυδίων του άνθρακα. Αυτές είναι, αυτή συγκεκριμένα η κατάργηση του άνθρακα, των εκπομπών άνθρακα, είναι σημαντική προτεραιότητα, όπως ξέρετε. Και η πρόταση της Κομισιόν προτείνει ότι 35% του προπολογισμού θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Είναι πολύ σημαντικό για τις μεταφορές, γιατί ξέρουμε ότι οι μεταφορές ε, συμβάλλουν πρέπει να συμβάλλουν, ιδιαίτερα στη μείωση των εκπομπών. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τους κλιματικούς στόχους, ούτω ώστε να παίξει πρωτοπόρο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθαρή ενέργεια και τα καθαρά καύσιμα. Αν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι ε, στις καθαρές μεταφορές, πρέπει να υπάρξει πολλή έρευνα και ανάπτυξη προς αυτήν την κατεύθυνση και ο Ορίζον Ευρώπη έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει προς αυτή την κατεύθυνση. Το νέο αυτό πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη συμπεριλαμβάνει τρεις πυλώνες. Οι μεταφορές είναι στο δεύτερο πυλώνα που είναι οι σφαιρικές προκλήσεις και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν τέσσερις τομείς θεμάτων, είμαστε στον τέταρτο ε, πακέτο θεμάτων. Αυτά είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, γι' αυτό στο σχέδιο γρομοδότησης προτείνω ότι ο πυλώνας 2 θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο, να είναι το 60%. Τώρα είναι γύρω στο 56% του συνολικού προϋπολογισμού για να υπάρξουν δυνατότητες για τη βιομηχανία μας να παίξει το ρόλο που πρέπει στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την κατάργηση των εκπομπών άνθρακα. Η Κομισιόν μοιάζει να έχει μειώσει λίγο την πρόταση για την χρηματοδότηση των μεταφορών, παρά το ότι συνολικά οι δαπάνε για έρευνα και ανάπτυξη έχουν αυξηθεί. Αν συμβάλλουμε, ε, αν εξετάσουμε λοιπόν συγκεκριμένα ποιε είναι οι χρηματοδοτήσεις για τις μεταφορές. Αλλά οι μεταφορές μπορούν και από άλλους τομεί θεμάτων, τα ψηφιακά για παράδειγμα, να χρηματοδοτηθούν. Και επίση και στον πυλώνα 3 υπάρχει το μέσο για τι μικρομεσαίες που παίζουν μεγάλο ρόλο στις μεταφορές. Άρα οι εταιρείε του τομέα των μεταφορών μπορούν, μπορούν και από εκεί να χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή να μην θεωρούμε ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από τον πυλώνα για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και την κινητικότητα μπορεί οι μεταφορές να χρηματοδοτηθούν και από άλλα τμήματα του Ορίζον Ευρώπη, ιδιαίτερα το τμήμα για την ψηφιοποίηση και από το τμήμα για τις μικρομεσαίες καλωσορίζω τη δυνατότητα για να υπάρξει έρευνα ε, ε, που συνδυάζει ε, τους διάφορους κλάδους και τις διάφορες επιστημονικές ειδικεύσει. Δεν θα πρέπει δηλαδή να περιορίσουμε τις χρηματοδοτήσεις σε κάποιους μόνο τομείς έρευνας, γιατί πολλές φορές η έρευνα και η καινοτομία συνδυάζει πολλούς τομείς. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ελαστικότητα μεταξύ των τριών αυτών πυλώνων. Πρέπει επίσης να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας. Για παράδειγμα, η... τα αυτόνομα οχήματα. Εδώ η εφαρμοσμένη έρευνα είναι πολύ σημαντική. Και, όπως ξέρετε, το χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ σφιχτό όταν εκπονούσα το σχέδιο γνωμοδότησης. Οπότε βεβαίως προσβλέπω και στη δική σας συμμετοχή, τις τροπολογίες σας και με χαρά θα συνεργαστούμε γιατί εξακολουθεί να είναι πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα στις επόμενες εβδομάδες. Αλλά κοιτάξτε, επειδή η πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ καλή, δεν έχουμε μεγάλες δυσχέρειες, τη συζήτησαν για χρόνια με τους εμπλεκόμενους φορείς και το Κοινοβούλιο συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Το κύριο μήνυμα θα πρέπει να είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην έρευνα και την καινοτομία. Ευχαριστώ κυρία Βρεκονέν. Πράγματι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Συμφωνώ απόλυτα. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την πρόταση και την εισηγήτρια για το σχέδιο νομοδότησης. Θέλω να παρακολουθήσουμε επικοδομητικά το θέμα αυτό, γιατί τα προβλήματα των μεταφορών στην Ευρώπη και στον κόσμο δεν θα τα λύσουμε αν δεν κάνουμε τεράστιες επενδύσεις στην έρευνα και χαιρετίζω ιδιαίτερα ότι εντός του πυλώνα σφαιρικές προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα αφιερώνουμε τα μεγάλα ποσά για το κλίμα, την ενέργεια και την κινητικότητα. Θέλουμε να αυξηθεί όμως η χρηματοδότηση συνολικά του προγράμματος αυτού. Οπωσδήποτε, επίσης, πρέπει να μειωθεί ε, η γραφειοκρατία όταν υποβάλλει κανεί αιτήσει και να μην χρειάζεται να κάνει δύο φορέ την ίδια δουλειά. Καλό είναι που το προτείνει η Κομισιόν. Το καθήκον μα ω Επιτροπή θα πρέπει να είναι μέσω τη γνωμοδότησή μα να επηρεάσουμε το επόμενο πρόγραμμα εργασιών διότι ένα πρόγραμμα έρευνας, εφόσον χρηματοδοτείται δημοσίως, πρέπει να έχει πολιτικές προτεραιότητες. Θέλουμε να υπάρχει καθαρή κινητικότητα που δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τα άτομα που ζουν στις ε, ε, μεγάλες πόλεις και στο κέντρο τους όπου υπάρχουν καλές συνδέσεις. Θέλουμε πιο ευφυείς μορφές κινητικότητας που να μην επιβαρύνουν τους χαμηλόμισθους. Πρέπει να έχουμε δικτυωμένα συστήματα ασφαλείας, όχι μόνο στο έδαφος, αλλά και στους ποταμούς και, τον, ε, και την αεροπορία. Δεν θα πρέπει να ε, καταργήσουμε δυνατότητες ατομικής μετακίνησης, αλλά να ενισχύσουμε τις ε, δημόσιες μεταφορές και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις διακοπές. Πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά χαίρομαι που θα συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους επικοδομητικά για να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταλόν, δεχτεί το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υποστηρίζουμε την αύξηση του προπολογισμού στα 97 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρότι θα θέλαμε παραϊσότερο, 120 θα προτιμούσαμε δις που θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε μειώνοντα το κοινό αγροτικό προπολογισμό. Επίση, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε ε, την ένταξη της κλιματικής διάστασης σε όλους τους τομείς. Ε, παρατηρούμε ότι με ε, τις καιρικές συνθήκες που επεκράθησαν στην Ευρώπη το τελευταίο καιρό δεν τηρούμε τους στόχους του προγράμματος. Οι προκλήσεις θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες στο μέλλον. Αυτό όμω αποτελεί και μια ευκαιρία για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και τι βιομηχανίε να διακριθούν εστιαζόμενε σε υψηλή ποιότητα κλιματικέ τεχνολογίε. Και εκεί έχουμε και κάποιε εξαγωγικέ δυνατότητε επιπλέον. Είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά το να δίνουμε χρήματα από το ορίζοντα Ευρώπη στη γεωγραφική βάση. Όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλου του σκοπού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε διαφορετικά ταμεία για διαφορετικού σκοπού. Πιστεύουμε ότι η αριστεία θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό κριτήριο στο οποίο θα ε, βασίζεται η επιλογή ενός έργου. Επίσης ανησυχούμε για τη ε, διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Εμείς ως νομοθέτες αφήνουμε πάρα πολλά ε, στην Κομισιόν όσον αφορά τις αποφάσεις. Εμείς ε, αναμένουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να βρούμε λύσεις για μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση με την εισηγήτρια, συγγνώμη. Επίσης πρέπει να εντάξουμε τη διάσταση του φύλου ε, στο όλο θέμα, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα στον τομέα τη έρευνα. Θα πρέπει οι γυναίκε να λαμβάνουν ίσε ευκαιρίες. Τέλο, πιστεύουμε επίση ότι το κομμάτι ε, των ψηφιακών ε, και της βιομηχανίας θα πρέπει να εστιάζονται περισσότερο στην ενέργεια, στις μεταφορές και στο κλίμα. Η βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, συμμετέχοντες σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θέλουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ενεργειακή απόδοση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νταλούντε. Κύριε Ρίκε, εκ μέρους της κυρίας Μάισνερ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Θα διαβάσω. Η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι προτεραιότητα του μελλοντικού προϋπολογισμού. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής. Η χρηματοδότηση που επενδύθηκε στην έρευνα και την καινοτομία φέρει τα μεγαλύτερα κέρδη. Η φιλόδοξη ατζέντα για την έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ευρώπης, αλλά και τις εταιρείες που θα πρέπει να δαπανίσουν, να επενδύσουν στην καινοτομία είναι ιδιαίτερη σημασίας το ζήτημα αυτό για να μπορέσουμε να καταφέρουμε το μέγιστο και να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η μόλυνση και η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας, καθώς και η μόλυνση των ωκεανών, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα ήθελα να επισημάνω την σημασία λοιπόν των αντίστοιχων ταμείων. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε εθνικό επίπεδο διάφορα προγράμματα όπως ε, την ε, αποφυγή της ρήπανσης των ωκεανών με πλαστικό θα πρέπει να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες που είναι όλο και πιο ενήμεροι σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται κοντά στους ε, πολίτες και στις ανησυχίες τους. Ευχαριστούμε κύριε Βίμ Βαντεκάμπα. Κυρία Γιάλα Σέντερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ την κυρία Βίρκουνεν για αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις. Και μια ερώτηση. Επειδή σήμερα το πρωί επειδή σήμερα το πρωί μας μίλησε για το συνδέοντα στην Ευρώπη. Γιατί λυπάμαι λιγάκι. Προτείνει ο ορίζον Ευρώπη να πάει από τα 94 δις γιατί είχε προτείνει ήδη σημαντική αύξηση του Κομισιόν, να πάει στο 131 δις. Εγώ να ρωτήσω πόσο είπατε να αυξηθεί το ΣΕΦ για τις μεταφορές ή για την ψηφιοποίηση. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι και με τον έλεγχο του προπολογισμού και εξετάζω από κάθε γωνία το ρίζο 2020. Νομίζω ότι μιλάμε για την έρευνα, λες και είναι το θαύμα του κόσμου και λέγονται απίστευτα πράγματα. Για παράδειγμα, η γεωγραφική κατανομή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς η συγκέντρωση, τα 10 σημαντικά προγράμματα με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που είναι. Δεν είναι ούτε στη δική σα, ε, ούτε στη δική μου χώρα, μόνο ένα και εν μέρη, από σπόντα. Γίνονται εκεί που υπάρχουν ε, μηχανικοί και εκεί που υπάρχουν κέντρα ε, έρευνας. Και δεύτερον, υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια και πολλά ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν με βάση το Horizon 2020. Πληρώνουν ε, ε, τους μισθούς των εργαζομένων και πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν ε, τους μισθούς των εργαζομένων τους από το Horizon 2020. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια και όχι απλώς να επιδοτούμε ε, επιχειρήσεις που μετά πουλάνε μετοχές. Δηλαδή, όταν λέμε να αυξήσουμε τόσο πολύ τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί, για ποιου, για πού, με τι έλεγχο και με τι αποτελέσματα. Γιατί πολύ συχνά η καινοτομία που είναι πώς περνάμε από την ε, βασική έρευνα στην ε, ε, ε, δημιουργία προϊόντων, πολλές φορές αποτυγχάνει και το ξέρουμε πολύ καλά. Και όταν αντιμετωπίζουμε βασικές ε, κοινωνικές προκλήσεις, ένταξη των ε, ε, μεταναστών, αντιμετώπιση της φτώχειας των ηλικιωμένων, αντιμετώπιση ανεργίας των νέων. Πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις του. Όταν προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις, δεν δίνουμε απαντήσεις. Σε τεχνικό επίπεδο, δεν λέω για πολιτικό επίπεδο, όπου να μην τα λέω. Θα έπρεπε λοιπόν, όταν κάνετε τόσο σημαντικές προτάσεις, τις οποίες χαιρετίζω, Καταπληκτικές προτάσεις. Και οι ερευνητές, όπως σας είπα, πάντα είναι καλοδεχούμενοι. Α, καμιά φορά όμως πρέπει να καταλαβαίνουμε με τι τρόπο αυτό το ορίζον Ευρώπη 21-27 θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κινητικότητας στην Ευρώπη. Και όχι απλώς να συνεχίσουμε να μοιράζουμε επιδοτήσεις ε, που ε, με πολύ χαρά τις δέχονται και ζουν πολλά χρόνια ε, από αυτές. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιν θέλει να προσθέσει κάτι. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. οι οποίε ε, να μην σχετίζονται άμεσα με το έγγραφο που μας παρουσίασε η κυρία Βερκούν, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένω να μου τις απαντήσει παρόλα αυτά. Γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι, πόσα ιδρύματα, πόσοι οργανισμοί ε, χρησιμοποιούν το Horizon 2020 ε, ή το Horizon Ευρώπη όπως ονομάζεται σήμερα, διότι έχω την εντύπωση ότι η ο μέσο ε, στον οποίο αναφερόμαστε απαιτεί ελάχιστη έρευνα και ότι πρακτικά ο τομέας των μεταφορών είναι κάπως ε, εκτός αυτού του θέματος. Δεύτερη ερώτηση, ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά, εμείς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούμε να απευθυνθούμε στο ορίζον Ευρώπη ή σε αυτό μπορούν να απευθυνθούν μόνο εξωτερικοί αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Είναι σαφές μετά αυτό που απαιτεί η DigiMove από το Horizon Ευρώπη ή δεν ζητάει τίποτα. Ήθελα να μάθω ποιοι θα είναι οι χρήστες. Και η τελευταία μου ερώτηση. Μήπως θα έπρεπε να πούμε ότι το Horizon Ευρώπη πρέπει να προβληθεί περισσότερο στον τομέα των μεταφορών. Ενδεχομένως όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Για παραδείγμα, και εκεί απαιτείται και άλλη έρευνα και αυτή θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Horizon Ευρώπη. Αυτά. Ευχαριστούμε. Κάποιες ερωτήσεις έτσι απευθύναν στην Κομισιόν. Δίνω το λόγο στην Κλάρα Ντελαρτόρ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκεστε εδώ. Ωραία. Καλώ ορίσατε στην Επιτροπή μα και ευχαριστούμε που θα συμβάλλετε και στη συζήτηση αυτή για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε στη συζήτηση αυτή και ευχαριστούμε και την εισηγήτρια η οποία κατάφερε με στενές χρονικά πλαίσια να ετοιμάσει την εισήγηση αυτή. Η μεταφορά, λοιπόν, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, ο τομέας των μεταφορών. Και είναι και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία, κατά το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις επιθυμίες της Κομισιόν να επενδύσουμε στην έρευνα. Το πρόγραμμα αυτό και συγκεκριμένα τομέας, ο τέταρτος τομέας, Πιστεύουμε εμείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτές την ανάγκη να, να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και όπως είπε και η εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση αυτά είναι ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τον τομέα των μεταφορών για την κινητικότητα που θα είναι στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι, όπως υπόθηκε. Και είναι ακριβώς αυτά τα ζητήματα που έθεσε και η εισηγήτρια που είχε στο μυαλό της και η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας. Βεβαίως θα πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλους τομείς, συγκεκριμένα με τον τομέα 3 σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η πρόταση της Επιτροπής έχει οθετήσει μια συστημική προσέγγιση για τις μεταφορές. Θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικά διάφορους τομείς για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το σύστημα στο σύνολό του και αυτό. Πολλές τροπολογίες τις οποίες η Κομισιόν θα ενσωματώσει με χαρά στο τελικό κείμενο γιατί θεωρούμε ότι βελτιώνουν την πρόταση. Αγαπητοί η συγγήτρια δεν θα επισέλθω στις τροπολογίες που αφορούν τον προϋπολογισμό, αλλά βεβαίως θα χαρούμε να στηρίξουμε ε, περαιτέρω επενδύσεις ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Πρώτα απ' όλα, έχουμε κάποιες τροπολογίες που αν ψηφιστούν μπορούν να ενσωματωθούν στην τελική μας πρόταση. Οι τροπολογίες 3 και 5 πιστεύουμε εμείς ότι αφορούν σε αυτό που είπε η, η την πρόθεση, την ενίσχυση των επενδύσεων. Επομένως, το πνεύμα της τροπολογίας αυτής που εμφανίζεται σε δύο-τρία διαφορετικά σημεία, θα χαρούμε να το εξετάσουμε μαζί σας. Υπάρχει μία τροπολογία που αναφέρεται συγκεκριμένα στον τομέα 3 και αφορά την ε, ψηφιακή βιομηχανία. Συμφωνούμε με το πνεύμα της τροπολογίας αυτής που μας υπενθυμίζει ε, την ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας την υποδομή και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουμε ότι έχουν πρόσβαση μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την τελευταία τροπολογία, τροπολογία νούμερο 9, συμφωνούμε, υπάρχουν ε, δύο διαφορετικά σημεία στην τροπολογία αυτή. Ένα από αυτά αναφέρεται στην ασφάλεια. Βεβαίω συμφωνούμε με την εισηγήτρια στην σημασία της ασφάλειας της μεταφοράς. Ε, θεωρούμε όμως ότι είναι καλύτερο να εξετάσουμε τις μεταφορές με έναν οριζόντιο τρόπο Πιστεύουμε λοιπόν ότι πολύ γρήγορα θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνούμε με α, το 35% του προϋπολογισμού που θα πρέπει μίνιμουμ να χρησιμοποιείται για την κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές ε, τις αποστολές, με συγχωρείτε, ναι, ισχύει αυτό που είπε η συγκήτρια, αλλά πιο συγκεκριμένα σε αποστολές κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τελευταίο θέμα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της γεωγραφικής διανομής των χρημάτων συμφωνούμε με την Επιτροπή. Τα επιδόματα θα πρέπει να δίνονται με βάση την αριστεία και τον αντίκτυπο και όχι με βάση την ε, γεωγραφική θέση. Αν θέλετε μπορώ να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, αν θέλετε μπορώ να το αφήσω για εργότερα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργειας, ερωτήματα που ακούστηκαν. Να κάνουμε ερωτήσεις και κύριε ε, Βίμ Βαντεκάμπα πώς μπορεί να ιτηθεί κάποιος ε, για αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να εστιαστούμε σε αυτά που ανισχούν εμάς ε, παρότι έχουμε μια γενικότερη εικόνα των πραγμάτων είμαστε ειδικοί της Επιτροπής Μεταφορών Έχετε απαντήσεις για αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ε, Δεν είχα καταλάβει καλά. Νόμιζα ότι η ερώτηση της κυρίας Αγιάλα ε, ήταν προς την εισηγήτρια για την αύξηση του προϋπολογισμού του διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να απαντήσω από αυτό, αλλά θα ήθελα να διαβεβαιώσω την κυρία Αγιάλα ότι εξετάζουμε στενά τη χρηματοδότηση του προγράμματος πλαισίου ε, βάσει των δικαιούχων που έχουν συμμετάσχει σε προσκλήσεις ε, ε, υποβολής προσφορών συγκεκριμένες και γνωστές σε όλους. Δεν εκπλήσει το ότι τα περισσότερα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας αφορούν περιοχές της Ευρώπης που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και στην καινοτομία. Πολλέ μελέτες, ε, το γνωρίζουν τα μέλη τη Επιτροπή αυτά, δείχνουν, αυτής ε, δείχνουν τη σχέση αιτία αποτελέσματος μεταξύ ε, της επένδυσης και της θωράξη των εθνικών συστημάτων έρευνα και καινοτομία, όπου τα διάφορα ταμεία, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, επικεντρώνονται σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται κάποια μέτρα, ώστε, ούτως ώστε όλα τα μέρη στην Ευρώπη να ε, έχουν κάποιο δυναμικό έρευνα και καινοτομία. Και όπως είπε και κάποιος άλλος ομιλητής, υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία πρώτα έχουν δημιουργηθεί για να αναπτυχθούν οι τοπικές και περιφερειακές ε, δεξιότητες σε έναν τομέα. Εμεί αυτό προσπαθούμε και σε αυτό έχει επικεντρωθεί το πρόγραμμα να έχουμε κάποια συνέργεια μεταξύ αυτού του προγράμματος και των άλλων προγραμμάτων του ΣΕΦ για να εφαρμοστούν ε, οι τεχνολογίες που έχουν οριμάσει, καθώς και τα προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να υπάρχει συνέργεια, ώστε η αριστεία να ευθυγραμμιστεί με τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης. Όσον αφορά το ποιο μπορεί να ετηθεί σε τέτοια προγράμματα, δεν θυμάμαι ακριβώ διατύπωση, αλλά θεωρητικά οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στο πρόγραμμα αυτό. Φυσικά εφόσον ε, τα προγράμματα παρουσιάζουν έχουν κάποια χαρακτηριστικά όπως κοινοπραξία, συνεργασία με ε, ε, τρία κράτη-μέλη τουλάχιστον. Ε, θεωρητικά όλοι μπορούν να αιτηθούν και οι δικαιούχοι από τρίτες χώρες δεν σημαίνει ότι θα λάβουν χρηματοδότηση, αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σα. Κυρία Βίρκονεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτον για τον προπολογισμό. Όπως ξέρουμε, το Κοινοβούλιο έλαβε μια απόφαση στην Ολομέλεια την Άνοιξη. Τι πρέπει να περιληφθεί στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο Είπαμε ότι ο προπολογισμό του ΣΕΦ πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τον τρέχοντα και το ότι το πρόγραμμα Horizon πρέπει να αυξηθεί για 50% και απλώς ε, ακολουθώ αυτή τη γραμμή. Γι' αυτό προτείνω 50% αύξηση. Σε τρέχουσες τιμές. Και γι' αυτό είναι 131 δις. Ο κύριος Νταλούντε είπε ότι θα πρέπει να είναι 120 δις αλλά νομίζω ότι εννοείται το ίδιο. Γιατί εσείς αναφέρεστε σε σταθερές και εγώ σε τρέχουσες τιμές. Ο προπολογισμό του ΣΕΦ είναι 42,7 νομίζω. 42,3 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Αλλά υπάρχει το νέο στοιχείο, η στρατιωτική κινητικότητα, άρα πώς θα ληφθεί υπόψη αλλά όπως ξέρετε αφορά και τις μεταφορές. Αλλά συζητάμε με τους συγητές και γι' αυτό. Για τον τομέα της ενέργειας και της ψηφιοποίησης έχουμε στην ουσία αυξήσει. Γι' αυτό δεν προτείνω αύξηση του προπολογισμού του ΣΕΦ. Γιατί αυτή νομίζω ότι ήταν η απόφαση του Κοινοβουλίου. Ο κύριος ε, Φαντεκάμπα για το πώς ε, κάνει κανείς αιτήσει για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη Κοιτάξτε, ε, όπως ξέρετε μόνο το 12% των αιτήσεων εγκρίνεται, άρα πρέπει να είναι πραγματικά κέντρα αριστείας ε, ε, όσοι αιτούνται. Και ε, ο τομέας των μεταφορών έχει λάβει πολλές χρηματοδοτήσεις, για παράδειγμα οι αερομεταφορές, το πρόγραμμα για το καθαρό αέρα ήταν ένα ευρύ πρόγραμμα και οι θαλάσσιες μεταφορές και οι αυτοκινητοβιομηχανίες ε, όλοι αυτοί ασχολούνται ιδιαίτερα με την έρευνα και ανάπτυξη και λαμβάνουν και κάποιες χρηματοδοτήσεις από το ορίζον 2020. Υπάρχουν δύο είδη χρηματοδοτήσεων για την θεμελιώδη έρευνα που διεξάγεται στα πανεπιστήμια, για θεμελιώδη λοιπόν έρευνα. Και κατόπιν ε, χρηματοδοτείται και η καινοτομία δηλαδή εκεί που είναι περίπου ήδη εμπορεύσιμα τα αποτελέσματα. Όλα αυτά έχουν επιτύχει πολύ, γιατί εδώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πολλές φορές ε, διοργανώνουν ομίλους μαζί με πόλεις, ερευνητές, επιχειρήσεις για θέματα, για παράδειγμα, αστικής κινητικότητας και για άλλες ε, καινοτομίες. Νομίζω λοιπόν ότι οι μεταφορές ήδη έχουν αξιοποιήσει ιδιαίτερα αυτούς τους πόρους και στο μέλλον νομίζω τα επόμενα χρόνια θα ασχοληθούμε και με, το, με την κλιματική αλλαγή που είναι κύρια προτεραιότητα ή μία από τις κύριες προτεραιότητες όπου έχει σημαντικό ρόλο να παίξει ο τομέας των μεταφορών. Πολλή έρευνα γίνεται επίσης και για την ενέργεια και χρηματοδοτείται και φυσικά και ψηφιοποίηση. Επίσης σημαντικό θέμα για τις μεταφορές. Λαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon. Οι μεταφορές ε, είναι λοιπόν σημαντικό και θα συνεχίσει να είναι και να αυξάνεται η σημασία του στα πλαίσια του προγράμματος αυτού στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Βίρκουνεν. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 3η 11 Σεπτεμβρίου. 11 το πρωί. Και να περάσουμε τώρα με την, ε, στη γνωμοδότηση προς την Μπούτζ για την ενδιάμεση έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο συγητής μας είναι ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ. Είμαστε λοιπόν στο 10. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρίκε που θα, παρουσιάσει, θα μας παρουσιάσει την περίφημη γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο μόλις αναφέρθηκε από την προηγούμενη συγγήτρια έχει ήδη υιοθετήσει δύο ψηφίσματα. Επαναλαμβάνω αυτά που υπόθηκαν. Δεν έλαβε θέση για διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων ε, το Connecting Europe Facility διότι σε αυτά τα ψηφίσματα υιοθέτησε κάποια αυξημένα νούμερα επί τριών σημείων το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη, το Erasmus και το COSME. Δεν ε, ανέφερε τίποτα για άλλα νούμερα. Δεν υιοθέτησε λοιπόν κάτι, δεν διόρθωσε τα νούμερα της Κομισιόν. Αυτό είναι σημαντικό για τα όσα θα πούμε στη συνέχεια, διότι στην πραγματικότητα το Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει θέση για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη στα ψηφίσματά του. Η έκθεση τώρα εδώ που έχουμε μπροστά μας λέει ότι κάθε επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες και τα αιτήματα της ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών για τον καθορισμό της οριστικής θέσης του Κοινοβουλίου σε θέματα προπολογισμού, σε θέματα πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή είναι η ε, έκθεση ε, Τη επιτροπή ω γνωμοδότηση για να καθορίσει budget την, τελευταία θέση του, την τελική θέση του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά ε, την Επιτροπή Μεταφορών, το θέμα είναι να υπογραμμίσουμε συγκεκριμένε προτεραιότητε, όχι να δώσουμε κάποια γνωμοδότηση για το σύνολο του δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσουμε ότι οι ανάγκε ε, σε εισαγωγικά ε, σε θέματα μεταφορών είναι αυξανόμενες δεδομένου ότι αυξάνεται, αυξάνονται οι μεταφορές, ε, ο αριθμός ανθρώπων και εμπορευμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιρροή στο περιβάλλον, ε, στις υποδομές, ε, θέτει θέματα ασφάλειας και οικονομικής απόδοσης. Ήθελα να επανέλθω σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, αναφερόμενο στο μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης. Εγώ είχα προτείνει μια τροπολογία για μεταφορά 20 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ από το ΦΕΝΤΕΡ ε, στο ΕΜΕΡ. Αλλά ήθελα να δώσω μια εξήγηση. Το, το ΕΜΕ δεν είναι ε, διάταξη για τα ευρωπαϊκά, διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, θέτει τα πράγματα υπό την άμεση διαχείριση της Κομισιόν. Να εξηγήσω, προηγουμένως είχαμε 10 δισεκατομμύρια ε, ευρώ τα οποία διαχειριζόταν ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υποδομών. Τα βάλαμε στο ΣΕΦ, μετά 10 δισεκατομμύρια τα βάλαμε στη... που... 10 δισεκατομμύρια που ήρθαν από τη συνοχή και επιπλέον 10 δισεκατομμύρια τα οποία τοποθετήθηκαν συνέχεια σε άλλα εργαλεία. Ουσιαστικά το ΣΕΦ δεν έχει φρέσκο χρήμα έχει 10 δισεκατομμύρια ευρώ που ε, έλαβε από τη συνοχή που θα πήγαινα για τις μεταφορές αλλά ε, δεν είχε προταθεί άμεσα και στην πρόταση που μας γίνεται δεν υπάρχουν χρήματα νέα. Ουσιαστικά έχουμε μειώσει τη δημοσιονομική προκοδότηση και όλοι λένε ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες, ο μηχανισμός λειτουργήσε πολύ καλά, θα έχουμε ένα πρόβλημα μη κάλυψη ε, των υποχρεώσεων από τις πιστώσει Οπότε η πρόταση που να πάρουμε 10 δισεκατομμύρια από την ανταγωνιστικότητα αυτό είναι πολύ λιγότερο από ό,τι είχαμε πάρει είχαμε κάνει προηγουμένως για τη συνοχή. Αυτό δεν δίνει νέους πόρους στις μεταφορές, διότι στην ανταγωνιστικότητα ήδη έχουν ε, δαπανηθεί πάνω από 5 για τις μεταφορές. Το να μεταφέρουμε λοιπόν απλά πόρους ε, από την ανταγωνιστικότητα στην άμεση διαχείριση ώστε αυτά που δαπανώνται για τη μεταφορά ε, να προσθέτουν αξία Έχουμε την υλοποίηση των ε, διευρωπαϊκών δικτύων και τα λοιπά. Ουσιαστικά το ΣΕΦ παραμένει ένα εργαλείο άμεσης διαχείρισης των πιστώσεων που ε, υπάρχουν για τις μεταφορές χωρίς να δημιουργούνται νέοι πόροι. Ε, ένα κομμάτι λοιπόν από την συνοχή και εγώ θα έλεγα και ένα κομμάτι από την ανταγωνιστικότητα. Δεν υπάρχει λόγος να τα αφήσουμε εκεί ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις. Όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μιλούσαμε για απόδοση των επενδύσεων στις μεταφορές όταν βρισκόνταν δεξιά και αριστερά και όταν τα συγκεντρώσαμε όλοι λέγανε ότι ήταν όλα καταπληκτικά. Λένε όλοι ότι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικές επενδύσεις, λειτουργήσαν πολύ καλά. Εγώ δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο τα κονδύλια ανταγωνιστικότητα του Φεντέρα που είναι πάνω από 80 ε, δισεκατομμύρια σε πληρωμές Αν δεν το πούμε εμείς, ξέρετε, δεν θα το πει κανένας. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει δεκτό, ακόμη και από την ίδια την Επιτροπή. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν. Να δώσουμε στην κυβέρνηση του Connecting Europe Facility επαρκή χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό δεν επηρεάζει το γενικό προπολογισμό. Δεν είναι επιπλέον πόρος αυτό που ζητάμε από τον προπολογισμό. Απλά μεταφέρουμε ένα κομμάτι από αυτά που έχουν δεσμευτεί για τις μεταφορές στην άμεση διαχείριση. Έτσι εξηγώ λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο φαίνεται λίγο παράλογο αλλά δεν είναι. Στην έκθεση θα προτείνουμε ε, να δημιουργηθεί και ένα κομμάτι για τον τουρισμό. Έχουν περάσει 18-12 χρόνια από τότε που έχουμε εντάξει τον τουρισμό ε, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη δημοσιονομικά. Αυτό είναι λίγο περίεργο, διότι είναι η μόνη ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αντιστοιχεί σε κανένα δημοσιονομικό κονδύλιο. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα για τους οργανισμούς, όπως ξέρετε, έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις σημαντικά, καθώς εντάσσουμε περισσότερες πολιτικές διακυβέρνησης. Αυτό ισχύει για την ΕΑΣΑ, για τον οργανισμό ναυτιλίας ε, κτλ. Οπότε πρέπει να προσέχουμε, δεν μπορούμε να τους δίνουμε όλο και περισσότερη δουλειά με την ίδια διακυβέρνηση και όσον αφορά τους ίδιους πόρους ε, ή μειώνοντας τους ίδιους πόρους. Τώρα για το... Ε, για το ΑΡΕΝΤΑ έχουμε σημαντικά προγράμματα. για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, και σίγουρα λοιπόν θα ακούσουμε και διάφορες παρατηρήσεις ε, για τις ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον προπολογισμό δεδομένων των προβλημάτων που τίθενται στον τομέα των μεταφορών. Αυτά κύριε Πρόεδρε είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία προτείνω εγώ θα έχουμε και όλες τις τροπολογίες ε, και από τη δική μας Επιτροπή και από την Επιτροπή Προπολογισμών φυσικά. Ευχαριστούμε. Αρχίζει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον Ντομίνικ Ρικέ για την ε, γνωμοδότησή του αλλά και για την εισαγωγή που μας έκανε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Είχαμε από το πρωί μία συνέλευση με την Ήτρε και την Τρανς και συζητήσαμε για κάποια από τα θέματα που έθιξε ο Ρίκε. Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2, γιατί ο Ντομινίκ μίλησε για την προοπτική επιστροφή στα νούμερα που είχαμε από το 2014-2020. Κάποια μέλη όμως ήθελαν υψηλότερα ποσά από το 12,3. Το 11,5 είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με τους συναδέλφους από τον τομέα της συνοχής. Το 12 δεν θα πρέπει να είναι ακόμη υψηλότερο. Είναι πολύ νωρίς για να αποφασίσουμε. Το 12,3 με συγχωρείτε. Τα 20 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμφωνώ, αλλά δεν θα είναι αυτό μια τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές μας ικανότητες, δυνατότητες. Γιατί με 20 δισεκατομμύρια, ουσιαστικά θα είχαμε στα χέρια μας 30 δισεκατομμύρια και θα είχαμε και έξτρα 20 δισεκατομμύρια. Μήπως μπορείτε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε τα νούμερα αυτά, τα ποσά αυτά. Και το τρίτο σημείο είναι ότι στην γνωμοδότηση δεν ε, αναφέρεται πουθενά η στρατιωτική κινητικότητα. Δεν είναι αναγκαίο πρώτα να καλύψουμε αυτό με δεδομένες τις συζητήσεις που είχαμε και σήμερα το πρωί. Γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Διαφορετικά, ο στρατιωτικός τομέας πραγματικά θα καταποντιζόταν από τον τομέα των μεταφορών. Κάποιοι θα έχουν διαφορετική άποψη, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Διαφορετικά μπορεί να καταλήξουμε να μην είμαστε αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την έρευνα τώρα με αρκετά προγράμματα όπως είναι το Clean Sky δεν θα θεωρηθούν κοινέ επιχειρήσεις και η Επιτροπή δείχνει να απομακρύνεται από την προοπτική. Μπορείτε να σχολιάσετε λίγο πάνω στο ζήτημα αυτό. Γιατί εμένα μου φαίνονται κοινέ επιχειρήσεις και θα πρέπει να συνεχίσουν ως τέτοιες. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Ευχαριστούμε κύριε Βαντεκάμπ. Κυρία Ντεμόντε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Έκανε μια πολύ πλήρη παρουσίαση. Έχουμε ένα εξαιρετικό σχέδιο γνωμοδότησης εδώ και ήθελα να τον συγχαρώ. Όσον αφορά το κομμάτι που αφορά τι μεταφορέ και τι υποδομέ, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε προτεραιότητα στι επενδύσει υποδομών και στι επενδύσει συντήρηση για να υπενθυμίσω δυστυχώ άλλη μια φορά το δυστύχημα που είχαμε στην Ιταλία, την κατάρρευση μιας γέφυρα. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ασφαλεία των πολιτών και για να δια, τους ε, διαβεβαιώσουμε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την ασφαλειά τους. Ο στόχο αυτός λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στο δημοσιονομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τα TNT, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα διασυνοριακά δίκτυα και στα missing links. Κυρίω για τα προγράμματα που έχουν ήδη ξεκινήσει από άψη χρηματοδοτική. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα να αναφέρεται το θέμα του τουρισμού, δηλαδή η ανάγκη να υπάρχει ένα ειδικό κονδύλι του προπολογισμού, αφού πρόκειται για τον τρίτο οικονομικό κλάδο στην Ευρώπη. Ο εισηγητής λοιπόν ε, ανέφερε πόσο επηρεάζει το ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αναφέρθηκε κάποιος οδηγός ε, για τα κονδύλια που δίδονται στον τουρισμό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει και μια γραμμή προπολογισμού ειδική για τον τουρισμό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, να αυξηθεί η ευελιξία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί και μια γρήγορη απάντηση ε, για τι απρόβλεπτε ανάγκε. Ε, εδώ βλέπουμε τι διάφορε ανάγκε που έχουν προκύψει λόγω τη μετανάστευση. Και τέλο, υπάρχει ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, το θέμα τη επαρκού επικοινωνία. Για να έχουμε ένα καλό μέλλον ε, ε, για τους ανθρώπους αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι η μετανάστευση αντιμετωπίζει διάφορα εμπόδια ε, και σήμερα βρίσκεται υπό επίθεση. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε μια θεσμική αναθεώρηση των συνθήκων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε και αποτελεσματική επικοινωνία προς τους πολίτες, διότι οι πολίτες ε, αισθάνονται ότι οι επιλογές τους δεν ε, γίνονται σεβαστές. Θεωρούν ότι υπάρχει μια πολιτική σε υψηλό επίπεδο που δεν δίνει πραγματικά απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά και σίγουρα και εγώ θα συμμετέχω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη βελτίωση αυτής της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ντεμόντε. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Λιβιέ Σιλά Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και όσους παρενέβησαν στο σημαντικό σημαντικότατο αυτό ζήτημα του προϋπολογισμού για τις μεταφορές σε ό,τι αφορά τα ποσά που αναφέρθηκαν υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες. Εμείς θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συγκρίνουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Τα νούμερα δεν είναι ενθαρρυντικά, αλλά αν κάνουμε την σύγκριση αυτή έχοντας υπόψη μας την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έχουμε μία αύξηση της τάξης του 4% και ένα σταθερό ποσό σε ό,τι αφορά την συνοχή. Και σε αυτό προστίθεται και το κομμάτι της στρατιωτικής κινητικότητας. Θεωρούμε ότι στο συνολικό πλαίσιο της πρότασης της Κομισιόν είναι μια ρεαλιστική πρόταση αυτή η οποία καταθέτουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΦΕΝΤΕΡ, Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι που να αναφέρεται στις μεταφορές για το Ταμείο της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εκεί ακολουθούνται οι προτεραιότητες που έχουν ήδη αποφασιστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρούσα πρόταση της Κομισιόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο αυτό για να στηρίξουμε ταμείο αυτό και ε, για να στηρίξουμε και τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Επομένως, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την δυνατότητα μιας γεωγραφικής εξέτασης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες που θα στηρίξει το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορούμε να δούμε αυτού του τύπου τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Πέρα από αυτό όμως, η πρότασή μας προβλέπει επίσης και τη δυνατότητα να μεταφερθούν με όριο το 5% για παράδειγμα να υπάρχει μια επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ των διαφόρων ταμείων κατά των ενδιαφερομένων κρατών μελών υπάρχει μια μικρή ευελιξία στον τομέα αυτό, κατά πέτηση των κρατών μελών που ενδιαφέρονται πάνω απ' όλα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την αναφορά που έγινε στα ρυθμιστικά όργανα και πιο συγκεκριμένα την ανάγκη ενός προεπολογισμού για τέτοιου τύπου όργανα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η πρόεδρος λέει ότι δίνουμε το λόγο και πάλι στον εισηγητή, στον κύριο Αγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές και θα εξετάσουμε πολύ ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες σας. Να σχολιάσω ότι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι ο φάκελός του είναι 380 δισεκατομμύρια και παίρνουμε 20 και τα θέτουμε υπό διαχείριση. Είναι ο ίδιος μηχανισμός και με τη συνοχή. Δεν τα αφαιρούμε, απλώς τα θέτουμε σε απευθείας διαχείριση. Άρα ίδιο όριο για το Ταμείο περιφερικής Ανάπτυξης και τον προπολογισμό. Τι μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα σχολιάσω στην ε, ελαστικότητα του 5% όπως δουν τα κράτη-μέλη δεν νομίζω ότι έχει αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι θα αξιοποιήσουν στα πλαίσια του τρέχοντος, της τρέχουσας διαχείρισης κάτι τέτοιο τα κράτη-μέλη. Αλλά κοιτάξτε, στον προηγούμενο προϋπολογισμό απαγορευόταν να να χρηματοδοτούνται οι μεταφορές στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας. για άλλες περιπτώσεις εκτός ανταγωνιστικότητας υπήρχε κάποια δυνατότητα. Αλλά βλέπουμε ότι τελικά ένα σημαντικό τμήμα της περιφερειακής ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε για τις μεταφορές. Αλλά πολύ λίγο ή καθόλου για προγράμματα που προσέθεταν αξία. Εγώ το ξέρω, ήμουν σε μία ε, γαλλική περιφέρεια. Δεν ξέρω τι τα κάναμε. Άρα το θέμα είναι εάν η διαχείριση των πόρων του Περιφερειακού Ταμείου από τα κράτη-μέλη για τις υποδομές μεταφορών τους επέτρεπαν να προσθέσουν ευρωπαϊκή αξία. Και να μην αναφερθώ σε αυτά που συνέβησαν ε, πρόσφατα για θέματα υποδομών και συντήρησης. Δεν μπορείτε να θεωρείτε και εκπλήσουμε που η Κομισιόν το θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται καλύτερα από την ίδια τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον τομέα των υποδομών. Και είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό ότι δίνουμε στην ε, συνοχή 10 δις με άμεση διαχείριση και όχι για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εξηγήστε μου γιατί. Ίσως ε, οι χώρες της συνοχής ε, δεν είναι αρκετά ικανές για να διαχειριστούν τους πόρους αυτούς προς το ευρωπαϊκό συμφέρον. Νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση αυτή που γίνεται, αλλά και θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει το Περιφερειακό Ταμείο να συμμετέχει στην προσπάθεια ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, δημιουργίας τέτοιας ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Κάνετε κάποιους υπολογισμούς ε, που βασίζονται στο ότι θα περάσουμε σε 27 από τις 28 χώρες. Άρα λέτε υπήρξε 4% αύξηση. Ναι. Αν υπολογίσουμε ότι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 15% επιστροφή, αλλά δεν το αξιοποιούσε πλήρω. Νομίζω ότι στην ουσία χάνουμε. Και θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε βέβαια τι σημαίνει τρέχουσες και τι σημαίνει σταθερές τιμές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Ντεμόντε για την συντήρηση και τις προτεραιότητες και με αυτό που είπε ο Βήμα για το στρατιωτικό και το πολιτικό. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαχείριση, αλλά ασχολούμαι μόνο με τις ε, ε αρχές. Καταλαβαίνω τι λένε οι συνάδελφοι για τις προτεραιότητες διαχείρισης, αλλά αυτό δεν είναι στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αφορούν άλλο κανονισμό αυτά όσο και αν συμμορίζουμε τις ανησυχίες σας, ε, δεν θα μπω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Πρέπει να εξακολουθήσετε να είστε τόσο αποφασισμένος και μαχητικός για να ε, στηρίξουμε τους στόχους μας. Προθεσμία για τις τροπολογίες 3η 11 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα. Οπότε λίγη δημόσια συνεδρίαση και θα συνεχιστεί η συζήτηση και κλεισμένο των θυρών για να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για να διακοπεί η μετάδοση μέσω ίντερνετ και να αποχωρήσει το κοινό. Φυσικά οι συνάδελφοι μπορούν να παραμείνουν. Δύο λεπτά παρακαλώ. Δύο λεπτά για να βγουν όσοι πρέπει να βγουν.